Um, λοιπόν, καλώς ήρθατε και πάλι. Ε, ζητώ συγγνώμη για την αλλαγή στο ωράριο, αλλά ήταν τόσο συναρπαστικά τα πράγματα στο ΕΚΟΦΗΝ ε, που ε, ο υπουργό κ. Σαρλή δεν μπορούσε να έρθει γιατί προείδρευε βεβαίω. Οπότε Αντιλαμβάνεστε πώς είναι τα πράγματα. Χαιρόμαστε όμως που ήρθε όπως μας είχε υποσχεθεί. Ε, να έρθει δηλαδή και να μας μιλήσει για τις ε, συστάσεις ε, αναχώρα τις οποίες αναφέραμε εντάχει στο Στρασβούργο. Τώρα όμως είναι πλέον επίσημες και αναμένουμε να ακούσουμε τι έχετε να πείτε και είμαι σίγουρος πως και οι βουλευτέ θα έχουν ε, κάποιες ερωτήσεις. Έχετε το λόγο. Thank you. Yes, indeed, it was quite pleasant to be uh, at the... Πράγματι ήταν μεγάλη ευχαριστήση μου να είμαι σήμερα στο Συμβούλιο. Πρώτη συνάντηση στην οποία προείδρευσα ήταν λοιπόν τιμή μου και προνόμιο να βρίσκομαι εκεί εκπροσωπώντας την Κύπρο. Βεβαίως Εκεί δεν εκπροσωπεί κανείς τη χώρα του, αλλά όλα τα κράτη-μέλη και τα 27 της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ήταν λοιπόν και ωραία συνάντηση και συναρπαστική. Πολλή δουλειά έχει γίνει ως τώρα. Ως προς το συγκεκριμένο θέμα, για το οποίο έχω προσκληθεί να, μιλήσω, στοιχεία για το ευρωπαϊκό Εξάμενο, δηλαδή, με μεγάλη χαρά να σας ανακοινώσω ότι σήμερα το Συμβούλιο Οικονομικών Υποθέσεων υιοθέτησε τις αναχώρα ειδικές συστάσεις. Ολοκληρώνοντας έτσι το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο του 2012. Περατώθηκε έτσι το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο του 2012. Η επίσημη έγκριση ακολουθεί την επίσημη έγκριση του Συμβουλίου στις 28 και 29 Ιουνίου. Οι δέσμοι συστάσεων συμπεριλαμβάνουν 27 ομάδες ειδικών συστάσεων αναχώρα για δημοσιονομικά μέτρα και οικονομικές μεταρρυθμίσεις. Αλλά και μια ομάδα συστάσεων για την Ευρωζώνη, την περιοχή της Ευρωζώνης. Όπως ξέρετε, αυτή είναι η δεύτερη φορά που το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο οργανώθηκε και φέτος συμπεριλάμβανε δύο νέα στοιχεία, δύο νέες ιδέες. Η πρώτη ήταν η αρχή της συμμόρφωσης ή εξήγησης, βάσει της οποίας το Συμβούλιο υιοθετεί τον εξής κανόνα. Να ακολουθεί τις συστάσεις της Επιτροπής ή δημοσίως να εξηγεί την θέση του. Αυτό ήταν πολύ, μια πολύ σημαντική προσθήκη. Επειδή διασφαλίζει μεγαλύτερη διαφάνεια και πάνω απ' όλα τη λογοδοσία για την όλη διαδικασία. Δεν θα ήταν υπερβολή να πούμε ότι αυτό επέτρεψε να ενδυναμωθεί η θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην όλη διαδικασία. Άλλωστε αυτή ήταν και η αρχική πρόθεση. Πέτυχε λοιπόν και μάλιστα τα πήγαμε και καλά. Το άλλο νέο στοιχείο ήταν η συμπερίληψη συστάσεων που προκύπτουν από τη διαδικασία διόρθωσης των μακροοικονομικών ανισορροπιών, MIP όπως λέγονται. Αφορούσαν 12 χώρες και έδειξαν ότι παρόλο που εκεί υπάρχουν ανισορροπίες, αυτές δεν είναι σε υπέρμετρο επίπεδο. Οι χώρες Αυτέ ήταν το Βέλγιο, η Βουλγαρία, η Κύπρο, η Δανία, η Ισπανία, η Φινλανδία, η Γαλλία, η Ουγγαρία, η Ιταλία, η Σουηδία, η Σλοβενία και το Ηνωμένο Βασίλειο. Αυτά τα δύο νέα στοιχεία επέτρεψαν η διαδικασία των συστάσεων να γίνει πληρέστερη από ό,τι του παρελθόν και λιγότερο περίπλοκη αφού υπήρχαν παράλληλες παράλληλοι σχηματισμοί του Συμβουλίου ταυτόχρονα. Επίσης εξετάστηκε το Σύμφωνο Ανάπτυξης και Σταθερότητας, καθώς και διαδικασία μακροοικονομικών ε, ανισορροπιών που ανέφερα και προηγουμένως, καθώς και γενικές διαφορετικές πολιτικές και για τα θέματα απασχόλησης, αυτά που αποφασίστηκαν από το Συμβούλιο Κοινωνικών Υποθέσεων. Ήταν αίσιο λοιπόν το πέρας των εργασιών μας σήμερα και είναι πλέον αρμοδιότητα των κρατών μελών να μεταφράσουν τις συστάσεις σε συγκεκριμένα μέτρα, δημοσιονομικά, διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις και ε, ωφέλη για την απασχόληση μέσω της νομοθεσίας τους. Λεπτομέρειες τώρα στο τι ζητήματα αφορούσαν κυρίω οι συζητήσει μα. Εάν δείτε τι λεπτομέρειε των συζητήσεων μεταξύ Συμβουλίου και Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την εφαρμογή τη αρχή ε, συμμόρφωση ή εξήγηση, δύο σημεία αξίζει να σχολιάσουμε. Πρώτον, ότι οι συζητήσει οδήγησαν σε κάποιες προσθήκε και αλλαγέ στις συστάσει με πλήρη συμφωνία και στήριξη τη Επιτροπή. Μάλιστα, για πολλά δεν ζητήθηκαν περαιτέρω αλλαγές στις συστάσεις τους, ενώ κατά δεύτερον, στις περιπτώσεις όπου δεν επετέφθη συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Συμβούλιο εξήγησε ακριβώς την στάση του. Η έκθεση με τις εξηγήσει αυτές εγκρίθηκε για αυτή επισήμω σήμερα και πολύ σύντομα θα λάβετε και αντίγραφο. Στην έκθεση Αξίζει να σημειωθεί ότι το επίκεντρο της συζήτησης και των αλλαγών αφορούσαν την αγορά της απασχόλησης, τις διευθυντικές αλλαγές και τα δημοσιονομικά. Λιγότερο για το χρηματοπιστωτικό τομέα. Συνολικά αλλαγές έγιναν και εξηγήσει δόθηκαν για συστάσεις σε 10 από τα 27 κράτη-μέλη. 27 χώρες. Σε 8 από τις 10 περιπτώσεις συμπεριλήφθησαν αλλαγές στις ε, συστάσεις για την απασχόληση και την αγορά εργασίας. 8 από τις 10. Η παρακολούθηση τώρα, η συνέχεια μάλλον του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου του 2012. Συνολικά, το Ευρωπαϊκό αυτό εξάμεινο έδωσε επιτυχή αποτελέσματα. Κατά δεύτερον, υπάρχουν τομεί όπου πρόοδο περαιτέρω πρόοδο μπορεί να επιτελεστεί, ιδίω λόγω των νέων στοιχείων τη διαδικασία. Μια τέτοια πρόκληση είναι να βρούμε την βέλτιστη χρήση του σύντομου χρονικού διαστήματος που έχουμε στη διάθεσή μας για συζητήσεις. Το ECOFIN σήμερα ξεκίνησε συζητήσεις για το πώς να βελτιωθεί το ίδιο το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο. Το σχετικό αυτό έργο θα προωθηθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τους αρμόδιους φορείς και θα τύχει εντελεχούς μελέτης από το ΕΚΟΦΗΝ του Οκτωβρίου, του ερχόμενου Οκτωβρίου. Εν ώψη όλων αυτών των στοιχείων, η Κυπριακή Προεδρία θα καλωσορίσει κάθε συνεισφορά του Κοινοβουλίου σχετικά. Η Κυπριακή Προεδρία παραμένει δεσμευμένη να προετοιμάσει ένα άριστο και εποφελές ευρωπαϊκό εξάμενο για το 2013. Αξίζει να σημειώσουμε από τη δική μας τη σκοπιά ότι το Συμβούλιο ενέκρινε σήμερα τα όσα ε, μπόρεσε να φέρει πέρα στο Ευρωπαϊκό Εξάμενο. Αυτά έχουν λήξει, έχουν περατωθεί σήμερα. Η όλη αυτή διαδικασία είχε και κάποιον αντίκτυπο. Δηλαδή, το Συμβούλιο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η αρχική κρατών και κυβερνήσεων φάνηκε ότι άσκησαν και επηρεάστηκαν από την όλη διαδικασία. Πριν από δέκα μέρες ήδη συζητήθηκε από τους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων το θέμα αυτό. Ένα άλλο σημαντικό στοιχείο είναι ότι οι διαδικασίες, οι κατάλληλες διαδικασίες έχουν πια εντοπιστεί, όπως προανέφερα, αναμένεται να επιτελεστεί εδώ βελτίωση, περαιτέρω βελτίωση. Όπως δήλωσα, βελτίωση περιμένουμε στον Οκτώβριο του 2012 και ως τότε θα οργανωθεί σύνοδος για την αναθεώρηση των διαδικασιών στο πλαίσιο που επίσης προανέφερα. Εάν το Κοινοβούλιο δηλαδή μπορεί να συνεισφέρει, αυτό θα ήταν ε, ευπρόσδεκτο. Σας ευχαριστώ. Thank Σας ευχαριστούμε κύριε Υπουργέ. Θα ακούσουμε τώρα τις ερωτήσεις των μελών της Επιτροπής. Πρώτα τους συντονιστές περιμένω, αλλά ε, δεν μου έχει κάνει νόημα. Θες το λόγο. Ε, όταν να μου προσφέρουν κάτι, Πολύ ευχαρίστω να το δεχτώ. Γιατί μερικές φορές ε, δεν λαμβάνω τίποτα. Συγγνώμη για την καθυστέρηση, γιατί δεν μπόρεσα παρά να ακούσω ένα μόνο τμήμα της παρέμβασης, αλλά σίγουρα το πιο ενδιαφέρον, εκεί που είπατε ότι ήσασταν έτοιμος να δεχτείτε τα στοιχεία και τις προτάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Εγώ με πιο νομικό τρόπο θα ήθελα να σας ρωτήσω πώς ε, προτίθεται η ε, Κυπριακή Προεδρία ή πώς αντιλαμβάνεται το ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε αυτή τη διαδικασία του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Γιατί θεωρούμε ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν είναι εδώ για να δίνει κάποια στοιχεία στην Προεδρία όταν έχουμε διάθεση και όταν είναι ωραίος καιρός. Έχουμε ένα πραγματικό, πραγματική εξουσία δημοκρατικού ελέγχου. Θεωρούμε ότι δεν θα κρίνουμε φυσικά κάθε χώρα, αυτό το κάνουν τα εθνικά κοινοβούλια, αλλά πιο γενικά πώς ε, θεωρεί η Προεδρία του Συμβουλίου ότι μπορεί να παίξει ρόλο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ποιος θα είναι αυτός ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και επίσης ποια είναι τα μέσα που θα διαθέσετε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να μπορεί να παρέμβει σε αυτή τη διαδικασία του εξαμήνου που είναι πάρα πολύ σημαντική για το μέλλον της οικονομικής μας ζώνης. Ευχαριστώ. Ο κύριος υπουργό θα απαντά την κάθε ερώτηση ξεχωριστά, έτσι για να μην τις ξεχάσω. Φυσικά, η Προεδρία του Συμβουλίου είναι η χώρα που εκπροσωπεί τις 27 χώρες μέλη. Και ως τέτοια, ως εκπρόσωπος, δίνει ε, γνώμες όχι της χώρας, ε, αλλά του Συμβουλίου ολόκληρου. Εμείς εκπροσωπούμε το Συμβούλιο. Δεν δίνουμε τις θέσεις της Κύπρου. Οπότε θα ήταν κάποιο, κάπως πρόωρο να λάβω θέση για το θέμα αυτό. Θα έλεγα πάντως, θα επαναλάβανα μάλλον αυτό που είπα και προηγουμένως. Δύο τινά δηλαδή. Πρώτον, όλοι θα συμβάλλουμε, γιατί μιλούμε για κάτι πολύ σημαντικό στην Ευρώπη. Οπότε όλοι έχουμε κάτι να προσφέρουμε και η συνεισφορά μπορεί να προέλθει από οποιοδήποτε με καλό πνεύμα και με σωστό τρόπο. Πάντως, η ερώτηση, κατάλαβα καλά, ήταν αν θα υπάρχει ένας νομικός, επίσημος, τυπικός τρόπος για ανάμειξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στη διαδικασία αυτή. Αλλά ακόμη βρισκόμαστε σε μια διαδικασία μάθησης κατά κάποιο τρόπο και από το πρίσμα του Συμβουλίου είχαμε μια πολύ σημαντική διαδικασία και είπαμε πρώτα να δούμε τι κάναμε, σήμερα το ολοκληρώσαμε, αλλά θα το επανεξετάσουμε, θα το αναθεωρήσουμε τον Οκτώβριο και με την εμπειρία που θα αποκομίσουμε θα συνδυάσουμε όλες αυτές τις εμπειρίες και φαντάζομαι τον Οκτώβριο θα είμαστε όλοι σοφότεροι προς όφελος των συμπολιτών μας των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οπότε έχουμε πολύ χρόνο μπροστά μας. Ας ακούσουμε, ας μάθουμε. Και η Προεδρία θα σημειώσει όλες αυτές τις πληροφορίες και θα τις θέσει προς συζήτηση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Νομίζω πως ίσως να είμαστε όλοι σοφότεροι βεβαίως τον Οκτώβριο γιατί η έκθεση της πρωτοβουλίας την οποία συντάσσει ο Ζαν επίσης κάποια στιγμή τον Οκτώβριο θα ψηφιστεί. Ναι, Ελίζα, ζήτησε το λόγο. Ευχαριστώ πάρα πολύ, θα μιλήσω αγγλικά. Ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε ξανά εδώ πέρα, κύριε Υπουργέ. Οι ερωτήσεις μου απευθύνονται προς το Συμβούλιο, όχι προς εσάς προσωπικά όχι προς ε, τον ε, εκπρόσωπο της Κύπρου, απλά προς το Συμβούλιο. Και έχω κάποιες ερωτήσεις. Πρώτα απ' όλα, ε, ήταν πάρα πολύ δραστήριο το Κοινοβούλιο όσον αφορά το πακέτο των έξι οδηγιών και βεβαίως δεχτήκαμε την ενίσχυση της Κομισιόν δηλαδή και την επιβολή ε, στα κράτη-μέλη, δηλαδή αυτό το comply or explain και ε, τι πρέπει να κάνετε αν δεν ακολουθείτε αυτές τις συστάσεις. Και η πρώτη μας ερώτηση είναι η ποιότητα αυτών των συστάσεων που δεν άλλαξαν. Και πάλι ξαναλέω, απευθύνομαι προς το Συμβούλιο, και προς εσάς. Η ασάφη, οι αδυναμίες είναι σαφείς. Είναι ασαφείς, είναι τα ίδια και τα ίδια, και η ίδια λυσίτα είναι μικρή ή μεγάλη χώρα, εξάγει ή όχι. Αυτό είναι το πρώτο σχόλιο. Και δεύτερον θεωρώ πως από το εξαπλό αυτό πακέτο ένα από τα σημεία προσθέμενης αξίας ήταν πως ζητήσαμε από την Κομισιόν να δούμε τι επιπτώσεις έχει κάτι το οποίο κάνει μια χώρα στις υπόλοιπες και αυτό αγνοήθηκε. Οπότε συνεχίζουμε ως συνήθως. Αυτό είναι το πρώτο μου σχόλιο. Δεύτερον, εάν δείτε τις αιτήσει εκθέσεις του Δουνουτού η αξιολόγηση του διεθνού Νομισματικού Ταμείου λέει για τη Γερμανία. Υπάρχουν οι όροι για μία ανάκαμψη η οποία θα οδηγηθεί από την ζήτηση στην μεγαλύτερη οικονομία της Ευρωζώνης μετά από μία περίοδο δημιουργίας θέσεων εργασίας. Θα υπάρξει λοιπόν μια φυσική αναπροσαρμογή τιμών και μισθών που θα πρέπει να αυξήσει τις εισαγωγές που σε ένα βαθμό θα αποκαταστήσουν την ισορροπία στην Ευρωζώνη. Στην δε βαθμολογία που είδαμε από την Κομισιόν οι χώρες του υπερβολικού ελλείμματος όπως και οι χώρες του υπερβολικού πλεονάσματος ε, θα πρέπει να θίγονται και οι δύο. Ε, γιατί υπήρχε ένα πλεόνασμα εμπορικό της Γερμανίας στις τάξης του 5,9 και το όριο ήταν 6% οπότε δεν μπαίνει υποπιτήρηση για ένα 0,1% αλλά κάποιες συστάσεις για την συνολική εσωτερική ζήτηση της Ευρωζώνης στη μεγαλύτερη οικονομία της η οποία έχει συσσωρεύσει πλεονάσματα ε, θα πρέπει να υπάρχουν στο κείμενο. Δεν υπάρχουν. Τρίτον, για τις χώρες υπό την επιτήρηση της ε, Τρόικας, η οποία, να μιλήσω για τη χώρα μου, Πορτογαλία, η οποία τα ακολουθεί όλα μέχρι κεραίας. Να δείτε το αποτέλεσμα, λέει, ακολουθήσαμε όλες τις ε, συστάσεις, δεν έχουμε ελληνικού στυλ ε, αμφιβολίες, τα έχουμε ακολουθήσει, αυξήθηκε το έλλειμμα, μειώθηκε η απασχόληση, χρεοκοπίες παντού και η σύσταση ποια είναι, συνεχίστε αυτή την πορεία. Ε, πότε δηλαδή αναμένουμε από το Συμβούλιο να δει τα αποτελέσματα αυτών των συστάσεων τελευταίο για την ε, εργασία. Όποιες συστάσεις και να κάνει ε, το Συμβούλιο, καθώς το κόστος της εργασίας φαίνεται πως είναι η μόνη μεταβλητή η οποία θίγεται εδώ πέρα, ε, να υπάρχει σεβασμός για τον κοινωνικό διάλογο, κάτι το οποίο είναι μια αρχή της Ευρωπαϊκής Δημοκρατίας και είναι περίεργο. Ε, εγώ σας ρώτησα, αλλά προφανώς δεν ήταν η κατάλληλη στιγμή. Όταν κάνετε συστάσεις προς την Ιταλία, ήταν εκεί πέρα η πρόταση της Κομισιόν που έλεγε πως το κόστος της εργασίας θα πρέπει να μειωθεί σε συνεννόηση με τους κοινωνικούς εταίρους και σύμφωνα με τις εθνικές πρακτικές. Αφού το εξέτασε το Συμβούλιο, αποφάσισε να διαγραφεί αυτή η πρόταση. Οπότε τώρα τι έχουμε? Να ενισχύσει την εφαρμογή του νέου μισθολογικού πλαισίου για να υπάρξει μια ευθυγράμμιση με την παραγωγικότητα κτλ. κτλ. Δεν υπάρχει δηλαδή διαβούλευση με τους κοινωνικούς εταίρους. Επιδείνωση. Παρ' όλα αυτά, όταν μιλάμε για τη Φιλανδία, η Κομισιόν, η Κομισιόν δεν είχε ζητήσει διαβούλευση των κοινωνικών εταίρων και λέει σεβόμενο πλήρω τον ρόλο των κοινωνικών εταίρων και των πρακτικές. Γιατί δύο μέτρα και δύο σταθμά. Αυτές είναι οι ερωτήσεις μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και ε, παραλαμβάνω αυτές είναι ερωτήσεις προς το Συμβούλιο, όχι προς σας προσωπικά. Ναι, το, το αντιλαμβάνομαι. Δεν ε, τι τίθεται ζήτημα προσωπικό. Θέσατε κάποια ζητήματα, αλλά βεβαίως πίσω από το κάθε ζήτημα και ερωτήσεις υπάρχει ένα στοιχείο ζητημάτων που, που ανέφερα. Μπορούμε δηλαδή να δούμε το καθένα από αυτά εις βάθος, να τα αναλύσουμε και να εκφράσουμε μια άποψη. Τι λέω εγώ, προτείνω κάποια, πως κάποια από τα σχόλια τα οποία κάνατε πράγματι έχουν κάποια αλήθεια και αυτό ακριβώς συνέβη σε αυτές τις αλλαγές. Έχει οριστεί μια ημερομηνία για να λάβουμε υπόψη όλα αυτά τα σχόλια τα οποία είναι πάρα πολύ χρήσιμα. Βεβαίως, όσοι να ήξερα πώς θα θέσετε αυτά τα ερωτήματα, έχω φέρει μαζί μου έναν έμπειρο γνώμονα επί της Γερμανίας, είναι και μισός Γερμανός και μελετάει αυτά τα ζητήματα εδώ και καιρό και είμαι σίγουρος πως θα μας διαφωτίσει για αυτά τα ζητήματα. Αλλά πριν δώσω το λόγο, σωστό αυτό το οποίο είπατε για την Πορτογαλία και αντιλαμβάνομαι την περιπλοκότητα γιατί και η δικιά μου χώρα την ίδια οδό θα ακολουθήσει. Προς τα εκεί οδεύει και η Κύπρος. Οι συνθήκες τώρα είναι τέτοιες ώστε το εξωτερικό περιβάλλον και όχι οπωσδήποτε τα εσωτερικά της χώρας μπορεί να οδηγήσει τις χώρες σε κατευθύνσεις οι οποίες δεν θα είχαν ποτέ ονειρευτεί. Και αυτό το οποίο έχουμε αυτή τη στιγμή είναι μια κατάσταση όπου έχουμε μια κρίση στην Ευρώπη και η μια χώρα επηρεάζει την άλλη. Κάποιες μικρότερες, κάποιες μεγαλύτερες. στην ε, δικιά μας την περίπτωση υπήρχε ένα πρόβλημα στην Ελλάδα και αυτό ε, επηρέασε και την Κύπρο και ενώ ε, επί σειρά ετών η οικονομία μας πήγαινε πάρα πολύ καλά τώρα βρεθήκαμε σε αυτή την κατάσταση οπότε το θέμα αυτό που θέσατε θα το θέσουμε και εμείς στους επόμενους μήνες και θα δούμε τι θα γίνει του επόμενου μήνε, ελπίζω όχι χρόνια, μέχρι να βρούμε την απάντηση. Τώρα δίνω το λόγο στον Αντρέα. Uh, Καλησπέρα σα. Είναι πολύ καλό να έχουμε αυτή την ενδιαφέρουσα συζήτηση με τα μέλη τη ε, Επιτροπή σα, του βουλευτέ και τι βουλευτέ, παρόλο που είναι μια δύσκολη συζήτηση για τι παρατηρήσει σα. Ξέρουμε όλοι ότι οι οικονομίε τείνουν να έχουν πολύ οι οικονομολόγοι μάλλον τείνουν να έχουν πολύ διαφορετικέ απόψει. Εγώ θα σα εκφράσω μια άποψη που θεωρώ ότι αποτελεί αντικείμενο συνένεση στο Συμβούλιο για αυτό που ρωτήσατε. Θα υπάρχουν βεβαίω και διαφορετικέ απόψει για παρόμοια ζητήματα και για το ίδιο ζήτημα. Τάσει τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η γενική αίσθηση είναι ότι είναι πιο συγκεκριμένε και δεσμευτικέ φέτο. Όμω σημειώνω αυτό που είπατε. Δηλαδή, νομίζω ε, εννοείται ότι πρέπει να πετύχουμε μεγαλύτερη πρόοδο προς την κατεύθυνση της εξειδίκευσης αναχώρα. Δηλαδή, να ορίζονται προτεραιότητες και ίσως τον επόμενο γύρο συζητήσεων να συμπεριληφθούν και χρονοδιαγράμματα εφαρμογής. Ως τώρα οι συστάσεις αυτές είναι αρκετά γενικόλογες. Δίνουν κάποια καθοδήγηση, αλλά όχι πολύ χειροπιαστή για την, για, τον καθημερινή, για την καθημερινή υλοποίηση των οικονομικών πολιτικών. Έπειτα ονομάσατε και εντοπίσατε το γεγονός ότι υπάρχει αλληλεπίδραση. Είναι πολύ δύσκολο να υπολογίσει κανείς τι συμβαίνει με αυτήν την αλληλεπίδραση μεταξύ των οικονομικών φαινομένων. Ξέρετε ότι αυτή τη στιγμή το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο επιχειρεί να μελετήσει αυτά τα φαινόμενα και δεν είναι πολύ απλό σε επίπεδο οικονομίας να πούμε ότι εδώ υπάρχουν αυτές οι ανισορροπίες, άρα αυτή η διαφορετική οργάνωση ή η ανάπτυξη. Όχι, εδώ χρειάζεται περισσότερη τεχνική μελέτη για να δούμε τέτοια φαινόμενα και να εξοικειωθούμε. Όμως σημειώνω την παρατήρησή σας. κατά την εξέταση των μεγαλύτερων ιδίως χωρών θα πρέπει να έχουμε υπόψη ποιε οι επιπτώσει των πολιτικών τους ε, για το σύνολο τη Ευρωζώνης και την Ευρωπαϊκή Ένωση βεβαίω. Αυτό είναι ένα σημείο που αφορά λόγω χάρη την Γερμανία, το σχολιάσατε. Εάν δει κανεί την βαθμολογία, το λεγόμενο scoreboard, είδαμε ότι υπάρχει προσέγγιση εξέτασης και των ελλημάτων στο ισοζύγιο πληρωμών και των πλεονασμάτων. Είπατε κι εσείς ότι και αυτό είναι σημαντικό, τα πλεονάσματα. Βέβαια είναι διαφορετικό το κέντρο βάρους, του, είναι διαφορετική βαρύτητα του θέματος αυτού. Και στο Συμβούλιο φάνηκε αυτό, είναι λιγότερο προβληματικό. Δεν μιλάω τώρα ως Κύπριος πολίτης, όπου έχουμε μεγάλες ανισορροπίες στο σημερινό ισοζύγιο αλλά έχει εντοπιστεί τέτοιο πρόβλημα. Ούτως ή άλλως. Γι' αυτό και μας απασχόλησε. Τώρα, για την Τρόικα. Η ουσία είναι ότι μαθαίνουμε. Μαθαίνουμε. Από την αρχή της διαδικασίας τα διδάγματα είναι διαρκώς μεταλλασσόμενα. Αυτή τη στιγμή τα προγράμματα έχουν περισσότερο στόχο την ανάπτυξη και όχι πλέον μόνο τα δημοσιονομικά μέτρα. Να απασχολεί η σειρά προτεραιοτήτων, η ατζέντα της ανάπτυξης, την οποία υπονοήσατε, και η διάσταση των τραπεζών. Ο χρηματοπιστωτικός δηλαδή τομέας θα πρέπει να καλύπτεται και θα αρχίσει να καλύπτεται είναι κάτι που λαμβάνεται σοβαρό υπόψη. Όμως ε, θα πρέπει και να κατανοούμε το εξής. Τα προγράμματα αυτά χρειάζονται χρόνο. Χρόνο για να δώσουν αποτελέσματα. Δεν είναι βεβαίως αυτό δικαιολογία. Κάποιες φορές και ο σχεδιασμός των προγραμμάτων πρέπει να βελτιώνεται, να είναι πιο σφαιρικά στο σχεδιασμό τους, αλλά νομίζω ότι η κατεύθυνση που έχει ακολουθήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι λίγο πολύ αυτή που περιέγραψα. Θα πρέπει παρόλα αυτά να δώσουμε χρόνο ώστε να μπορέσουμε να δρέψουμε τους καρπούς των προσπαθειών μας. Ξέρετε ότι η όλη απόπειρα είναι δυσχερής. Και μιλώντας και υπό την ιδιότητα του Κυπρίου πολίτη, αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε και εμείς που επιτήρησε σε πρόγραμμα. Το άμεσο μέλλον για μας θα περιέχει ένα σωρό προκλήσεις και από οικονομικής και κοινωνικής και πολιτικής άποψης, σε επίπεδο και της οικονομίας. Εδώ τώρα για τις ειδικέ συστάσεις ε, για την Φιλανδία και την Ιταλία, προφανώς οι δύο χώρες δεν είναι παρόμοιες. Δεν θέλω εδώ να τοποθετηθώ, διότι δεν έχω εξειδικευμένες γνώσεις. Βεβαίως, αναγνωρίζει κανείς εύκολα ότι η περίπτωση της Ιταλίας με τα προβλήματα ανταγωνιστικότητας δεν προσωμιάζει με αυτή της Φινλανδίας. Ίσως η διαφοροποίηση να προκύπτει και από αυτό που σωστά αναφέρατε στην αρχή της παρέμβασής σας. Οι χώρες που είναι διαφορετικές θα πρέπει να καλύπτονται και με διαφορετικές συστάσεις. Σας ευχαριστώ. Ο Όλε από τους φιλελεύθερους. Ευχαριστώ. Κύριε Υπουργέ, Έχω κανένα δύο ερωτήσεις, μερικές γενικές και άλλες πιο ειδικέ. Διαρωτώ με πώς προχωρεί η συζήτηση, γιατί έχουμε τις συστάσεις, γίνονται κάποιες αλλαγές φαντάζομαι σε αυτές και ίσως και γίνονται κάποιες αλλαγές στις τελευταίες στιγμής κιόλας στις συστάσεις. Τι ακριβώς συμβαίνει και για ποιο λόγο. Αυτό θα ήταν πολύ ενδιαφέρον. Είναι ανοιχτή συζήτηση ε, ή μήπως όλα έχουν προκαθοριστεί. Η μηπω ολα εχουν προκαθοριστει η βουλγαρια και η Μάλτα ψήφισαν κατά. Για ποιο λόγο και ποιες είναι οι συστάσεις που δεν δέχτηκαν οι δύο αυτές χώρες. Η δική μου πατρίδα, η Σουηδία, ε, και η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, λέει ενθαρρύνει αυξημένη ελαστικότητα στους μισθούς. Αλλά αυτές ε, οι λέξεις έχουν διαγραφεί από τις ε, συστάσεις του Συμβουλίου και συζητήθηκαν ε, διεξοδικά στην Σουηδία. Φαντάζεστε γιατί. Και έχω και δύο επιπλέον ερωτήσεις. Ο κύριος Μπόργκ, ο Υπουργός Οικονομικών της Σουηδίας, ο συνάδελφός σας, είπε το Σαββατοκύριακο ότι η Ελλάδα είναι σχεδόν σίγουρα ότι θα χρεοκοπήσει. Ποια είναι η δική σας γνώμη. Και ο Φιλανδός ο Υπουργός Οικονομικών είπε αυτό το Σαββατοκυριακό πολύ έντονο βλέπετε στη Σκανδιναβία ότι η Φιλανδία μπορεί να εγκαταλείψει και το ευρώ αν κληθεί να πληρώσει για τις χώρες του Νότου και για να σωθεί το ευρώ. Αυτές ήταν οι ερωτήσεις μου. Σας ευχαριστώ. Uh, θα προσπαθήσω πάλι να απαντήσω με τη βοήθεια και του συναδέλφου του παρακαθημένου. Να ασχοληθώ με τα δύο πρώτα θέματα που θίξατε. Ε, δεν νομίζω ότι είναι δόκιμο να σχολιάζουμε δηλώσεις άλλων. Πάντως το θέμα είναι πολύ σημαντικό και μας αφορά και μας προβληματίζει, γι' αυτό και θα κάνω ένα σχόλιο. Δεν έχει νόημα ποιο το είπε ή με ποιο τρόπο. Θα μπορούσε να, θα μπορούσε να το είχε πει και σε άλλο πλαίσιο ή να ήταν διαφορετικά τα συμφρασόμενα. Πάντω η κατάσταση στην Ελλάδα είναι όντω πάρα πολύ σοβαρή. Το είπα και εγώ ότι τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η δική μου πατρίδα, η Κύπρος αυτή τη στιγμή, δεν προέρχονται από την οικονομία της ε, δικής μου πατρίδας, αλλά είναι συνέπειες της ε, οικονομικής κρίσης της Ελλάδας και αυτή η κρίση, αυτή η αποτυχία ουσιαστικά η οικονομική της Ελλάδας προκάλεσε και τα προβλήματα της Κύπρου. Και στις αρχές του χρόνου αποφασίστηκε να γίνει ένα κούρεμα των ελληνικών ομολόγων και είχαμε και το PSI, με το PSI. Και ήταν τεράστιο το κόστος αυτό. Ε, για τις δικές μας τράπεζες που είχαν επενδύσει, ήταν ιδιαίτερα εκτεθειμένες σε ελληνικά ομόλογα. Οι τράπεζες μας στην Κύπρο είχαν ε, επενδύσει και ανοίγοντας και θηγατρικές. Αλλού και εξαιτία του κουρέματος βρέθηκα σε πολύ δύσκολη θέση. Αν μια χώρα ε, έχει μια οικονομία σε τόσο δεινή κατάσταση, τι γίνεται. Και αυτό είναι το ερώτημα που μας προβληματίζει αυτές τις μέρες. Έγινε λόγος για μια τραπεζική ένωση. Γίνεται λόγος για μια ενιαία υποπτική αρχή στην Ευρώπη, ώστε να ελεγχθούν τέτοιου καταστάσεις. Γιατί πιστεύω ότι αν υπήρχε μια τέτοια ενιαία εποπτική αρχή στην Ευρώπη πριν από δέκα χρόνια, τουλάχιστον. Είμαι βέβαιος ότι σήμερα δεν θα είχαμε αυτά τα προβλήματα. Αλλά τα αντιμετωπίζουμε, η πραγματικότητα είναι αυτή, δεν μπορούμε να τα αποφύγουμε, θα πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε, ούτε μπορούμε να εθελοτυφλούμε. Και ε, μία σαν το μόνιμο μηχανισμό στήριξης και το μηχανισμό χρηματοπιστωτικής σταθερότητας δημιουργήθηκαν. Και ο στόχος τους είναι, χωρίς να βλάψουν τα υπόλοιπα κράτη της Ευρώπης να μπορέσουν να επιλύσουν τέτοιου είδους θέματα που είναι χρηματοπιστωτικά. Πριν από πολλά χρόνια, όταν είχα έρθει πάλι εδώ στο Κοινοβούλιο, στο Στρασβούργο ήταν τότε, είχα πει ότι χαίρομαι ιδιαίτερος και αισθάνομαι ιδιαίτερη τιμή και προνόμιο που βρίσκομαι ενώπιόν σας. γιατί ε, είναι ευχάριστο που όλες αυτές οι χώρες κάθονται στην τράπεζα των διαπραγματεύσεων, συζητούν και παρά τη δύσκολη κατάσταση καταλήγουν σε λύση. Συνήθως η λύση δεν εμφανίζεται από την αρχή. Μπορεί να προκύψει ένα μήνα μετά, ένα χρόνο μετά, μπορεί και μια διετία μετά. Πάντως αργά ή γρήγορα, με ειρηνικό τρόπο και με πολύ πολιτισμένο τρόπο, καταφέρουμε να βρούμε λύση στα προβλήματα. Θα θυμάστε ότι τον περασμένο αιώνα τα πράγματα ήταν πολύ διαφορετικά. Δεν είχαμε αυτό το προνόμιο. Γι' αυτό είπα ακριβώ ότι είναι τιμή για μένα και είναι προνόμιο που ζω σε αυτή την εποχή. Αλλά δεν έχουμε επιλύσει ακόμη όλα τα προβλήματα. Τα προβλήματα υπάρχουν ακόμη και με πνεύμα συνεργασίας θα πρέπει να καταφέρουμε να τα επιλύσουμε. Επαναλαμβάνω, είναι ιδιαίτερα επώδυνη αυτή η κατάσταση και για μένα, γιατί η πατρίδα μου παρόλο που είχε καλή οικονομία, τελικά έχει πληγεί από αυτήν την αλληλεπίδραση, αυτή τη μετάδοση του προβλήματος από άλλη χώρα. Ελπίζω πάντως, πραγματικά ελπίζω, ότι τελικά με αλληλεγγύη και από τους συμπολίτες των άλλων χωρών θα καταφέρουμε να βρούμε λύση, ώστε να μην έχουμε μια χώρα σαν την Ελλάδα με μια πραγματικά αποτυχημένη οικονομία. Γιατί αν η οικονομία μιας χώρας καταρρεύσει, σήμερα είναι η Ελλάδα, μπορεί άλλη, μέρα, άλλη φορά να είναι άλλη μέρα, η αλληλεπίδραση, το αποτέλεσμα, το αρνητικό μπορεί να μεταδοθεί και στην υπόλοιπη Ευρώπη. Δεν θέλουμε τέτοια αποτυχία, θέλουμε να αποτρέψουμε κάτι τέτοιο. Βέβαια, το προνόμιο της συμμετοχής στην Ευρωπαϊκή Ένωση συνεπιφέρει και κάποιες ευθύνες. Η Ελλάδα έχει ευθύνες και θα πρέπει να τηρήσει τις υποχρεώσεις της, της να αναλάβει τις ευθύνες της, αν θέλει να δεχτεί την αλληλεγγύη από τους υπόλοιπους εταίρους της. Νομίζω ότι αναφέρθηκα κάπως γενικά στα δύο θέματα. Τα πρώτα, στα δύο τελευταία θέματα, μάλλον θα δώσω το λόγο στον Ανδρέα για τα υπόλοιπα. Ε, I think... Νομίζω ότι πράγματι θίξατε ένα ζήτημα σοβαρότατο, πολιτικού και τεχνικού διαλόγου για τις συστάσεις. Ξέρουμε ότι το όλο πλαίσιο του διαλόγου πρέπει να βελτιωθεί. Αυτή τη στιγμή η διαδικασία προβλέπει ότι ξεκινάει όλη αυτή η προσπάθεια από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι χώρες έχουν τη δυνατότητα να συζητήσουν σε περισσότερο διμερές βέβαια επίπεδο με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Κάποιες χώρες ακολουθούν διαφορετικές πρακτικές, άλλοι έχουν και συμμετοχή κοινωνικών εταίρων ή των κοινοβουλίων τους με τρόπο πρακτικό κιόλας σε κάποιες χώρες υπάρχουν ε, άλλες πρακτικές. Τα στοιχεία αυτά θα πρέπει να ληφθούν υπόψη. Χρειαζόμαστε περισσότερο χρόνο. Είναι σαφές ότι οι συζητήσεις ολοκληρώνονται πολύ σύντομα και αυτό δεν επιτρέπει λεπτομερείς ε, συζητήσεις για τα διάφορα θέματα. Και τώρα για να περάσω στις λεπτομέρειες, τις συγκεκριμένες ερωτήσεις για την Μάλτα και τη Βουλγαρία εδώ αυτά δεν έχουν να κάνουν με τις ε, χώρες και τα ιδιαίτερα προβλήματα τους. Αυτό που πρέπει να σκεφτούμε είναι ότι αυτή τη στιγμή τα χρονικά περιθώρια είναι σημαντικά γιατί και είναι δύσκολη. Θα πρέπει να σκεφτούμε και το αύριο. Όμως θα πρέπει να εξοικονομήσουμε χρόνο και να συζητήσουμε προβλήματα για τα ανεπιλήτα θέματα της Βουλγαρίας και της Μάλτας. λόγω χάρη για το ποιο είναι ο πολιτικός, οικονομικός, κοινωνικός αντίκτυπος ε, των αλλαγών ε, στο, στις συντάξεις και τα επιδόματα ή το κόστος του βιωτικού, του, της ζωής στις δύο χώρες αυτές. Ευχαριστώ, Σβέν. Ναι. Θα ξεκινήσω στα γερμανικά και μετά θα κάνω και μια ερώτηση στα αγγλικά. Πρώτα απ' όλα, σας καλωσορίζω και εγώ στην Επιτροπή μας ξανά. Κατά την άποψή μου, έχοντας δει τις προτάσεις Κομισιόν και το τι αποφασίστηκε, οπωσδήποτε υπάρχει μία πρόοδος. Βλέπουμε πως ε, Υπάρχουν κάποια όρια στο έρωμα αυτής της πρότασης. Είχαμε κάποιες απόπειρες να αποδυναμωθεί, αλλά συνολικά έχει διατηρηθεί ο πυρήνας. Γιατί θα θυμάστε πως κάποιε κάποιες χώρες δεν έκαναν καθόλου καμία αλλαγή. Οπότε αυτό είναι θετικό και δείχνει και τον ενισχυμένο ρόλο της Κομισιόν όπως είπατε. Η χώρα όπου εγώ, ε, την οποία εγώ γνωρίζω καλύτερα, τη Γερμανία, τη δική μου, ε, για αυτήν πρέπει να πούμε πως έχουμε την εντύπωση πως το Συμβούλιο βρήκε ένα νέο κόλπο για να μην πάρουν την υπόθεση στα σοβαρά. Πρώτα απ' όλα η σύσταση είναι ισορροπημένη. Δεν μπορούμε να πούμε πως ε, θα γίνουν όλοι ξαφνικά ε, φιλελεύθεροι και πως μόνο μπορούν να μειώνονται οι μισθοί λέει πως πρέπει να αυξηθούν οι μισθοί ανάλογα με την παραγωγικότητα, πως πρέπει να επενδυθούν περισσότερα στην εκπαίδευση, στην έρευνα, πως δεν εξυπηρετεί αρκετά τους ασθενέστερους το σύστημα εκπαίδευσης, πως πρέπει να απελευθερωθούν κάποιες υπηρεσίες όπου είναι δύσκολη η πρόσβαση στην αγορά. Α, έχει φύγει και ο Βολφ Κλίντς. Ε, φορούν κάποιοι πελάτες του, τους ε, ψηφοφόρους του, με συγχωρείτε, φαρμακοποιούς ε, και τα παρόμοια και ζητάνε μάλιστα να αλλάξουν τα φορολογικά κίνητρα στον τομέα α, των, της φορολόγησης των οικογενειών όπου εργάζονται και οι δύο. Η Γερμανία δεν ζήτησε κάποια αλλαγή. Αν δει κάποιος βεβαίως λεπτομέρειες βλέπουμε πως οι συστάσεις είναι λίγο πολύ ίδιες με πέρσι. Γιατί δεν ακολουθούθηκαν οι συστάσεις. Και άρα τίθεται το ερώτημα, τι γίνεται ε, στην περίπτωση που δεν αλλάζουν οι συστάσεις, όπου οι χώρες λένε δεν κάνουμε τίποτε. Δεν υπάρχει εδώ πέρα comply or explain. Δηλαδή, αν οι χώρες απλά τα αγνοούν αυτά, εμφανίζονται σε ένα πίνακα, λένε εν μέρος ε, το ακολούθησαν και μιλάμε για κάτι λεπτομέρειες, έτσι εν μέρη το ακολούθησαν, αλλά θα ήθελα να μας πει το Συμβούλιο τι σκοπεύει να κάνει με χώρες όπου επί σειρά ετών έχουμε τις ίδιες συστάσεις ξανά και ξανά και θέλω να μας πει και η Κομισιόν. Τι σκοπεύει να κάνει με τις χώρες που λένε «Ωχ, δεν μας παρατάνε και αυτοί, πας ε, λένε εκεί πέρα ό,τι θένε, ποιο του δίνει σημασία». Και τέλος μια παρατήρηση στα αγγλικά. Αναφέρατε την ανάγκη να υπάρξει αλληλεγγύη προς την Κύπρο και προκειμένου να ξεπεραστούν προβλήματα που οφείλονται στην αλληλεπίδραση και την μετάδοση των προβλημάτων της Ελλάδας. Βλέπουμε πόσο κρίσιμη είναι η κατάσταση στην Κύπρο. Νομίζω ότι σε ευρωπαϊκό επίπεδο πραγματικά θα πρέπει να επιδειχθεί η αλληλεγγύη για να μην καταρρεύσει το τραπεζικό σύστημα. Όμως ταυτόχρονα διαρωτώ Η αλληλεγγύη είναι μονόδρομος Συζητήσαμε το φορολογικό σας σύστημα ήδη μια φορά στο Στρασβούργο. Επιτρέπει την εισρωή ε, μερισμάτων με μηδενικά τόκια και την εκροή. Γι' αυτό 250.000 ε, εταιρείε έχουν το δυνατό τους στην Κύπρο. Όχι γιατί λειτουργούν μέσα στην τοπική οικονομία, αλλά γιατί μάλλον είναι πολύ ευνοϊκό το φορολογικό σας περιβάλλον. Διερωτώ με λοιπόν, εάν ζητάτε στήριξη από τα ευρωπαϊκά συστήματα και τους ευρωπαϊκούς μηχανισμούς, θα μπορούσατε να αλλάξετε το σχεδιασμό του φορολογικού συστήματος ώστε να μην γίνεται αντικείμενο εκμετάλλευση ώστε κάποιοι να αποφεύγουν τη φορολόγηση αλλού. Νομίζω ότι αυτό θα ήταν δίκαιο εφόσον ζητάτε επίδειξη αλληλεγγύης απαντήσω στο τελευταίο ερώτημα και πάλι πρώτο. Η αλληλεγγύη στην οποία αναφέρθηκα δεν αφορούσε την Κύπρο, αλλά γενικότερα την κατάσταση. Η Ελλάδα είναι η χώρα στην οποία γεννήθηκε και προέκυψε το πρόβλημα. Η μετάδοση αυτή, η λεπίδραση του προβλήματος επηρέασε την Κύπρο. Πιστεύω λοιπόν ιδιαίτερο στην έννοια της αλληλεγγύης και εννοώ με αυτό ότι όπως και οι Έλληνες περιμένουν αλληλεγγύη από τους άλλους, θα πρέπει να λάβουν πολύ σοβαρά υπόψη και τις υποχρεώσεις που έχουν αναλάβει προς την Ευρώπη. Αυτό εννοούσα και για την Κύπρο. Όμως, η έννοια της αλληλεγγύης μπορεί να αφορά την οποιαδήποτε χώρα βεβαίως. Θα μπορούσε να ισχύει για οποιαδήποτε χώρα. Αυτό είπα. Πιο συγκεκριμένα σε κάτι που αναφέρατε νωρίτερα δεν θα μιλήσω για το φορολογικό σύστημα. Νομίζω ο σκοπό τη συνάντηση αυτή δεν ήταν να μιλήσουμε για την φορολογία. Αν όμω κάποιο έχει τέτοιε πληροφορίε, ε, γιατί εγώ πιστεύω ότι οι πληροφορίε που έχετε δεν είναι ακριβεί, αν ε, έχετε συγκεκριμένε πληροφορίε θα σα απαντήσω γραπτό. Διότι φαίνεται ότι κάποιοι θέλουν να θέτουν ξανά και ξανά το ζήτημα τη φορολογία στην Κύπρο. Είναι πολύ χαμηλοί φορολογικοί συντελεστέ στην Κύπρο και αυτό ισχύει για όλου και για του ντόπιου για τον οποιονδήποτε Ευρωπαίο, για οποιονδήποτε πολίτη του κόσμου που θέλει να έχει επιχειρηματική δραστηριότητα στην ε, Κύπρο. Είναι μια χώρα με σχεδόν μηδενικό φόρο. Οι συστάσεις χώρα τώρα και το κατά πόσον λαμβάνονται υπόψη ή όχι. Είπατε ότι κάθε χρόνο οι συστάσεις είναι λίγο πολύ ίδιες. Έχετε δίκιο. Όμως αυτός είναι ο λόγος που η... ανέφερα ξανά και ξανά την αρχή αυτή το συμμόρφωση ή εξήγηση. Comply or explain. Είναι τώρα ευθύνη του Συμβουλίου. Αυτή την σύσταση, αυτή την αρχή να φροντίσει να την υλοποιήσει. Το Συμβούλιο έχει αναλάβει τεράστια ευθύνη που προηγουμένως δεν υπήρχε. Εφ' εξής, και αυτή είναι η ομορφιά της όλης διαδικασίας, το σύστημα, αυτή, το σύστημα αυτό εξελίσσεται αργά μεν, αλλά με αποτελεσματικό τρόπο. Το Συμβούλιο αναλαμβάνει πλέον ευθύνη εξήγηση. Για δύο συνεχόμενα χρόνια, α πούμε ότι κάποιο έχει την ίδια σύσταση. Άρα, ναι, η παρατήρησή σας μπορεί να είναι σωστή, όμως εγώ ελπίζω και πιστεύω ότι ο μηχανισμός που ακριβώς τώρα προβλέφτηκε θα αρχίσει να αποδίδει αποτελέσματα πολύ σύντομα. Και πάλι θα απαντήσει και ο συνάδελφος, ο παρακαθήμενος μάλλον, Ναι, ε. λοιπόν, έχουμε ακόμα 8 συναδέλφους περιμένουν να κάνουν καμία ερώτηση. Η πτήση μου εμένα φεύγει τα μεσάνυχτα, οπότε είμαι στη διάθεσή σας. Ε, κοιτάξτε, λέει πρόεδρος, κάποιος άλλος θα αναλάβει την ε, προεδρία. Λοιπόν, και η κατόπιν για το ECR. Όχι, εγώ θα είμαι σύντομη γιατί θεωρώ πως είχαμε ήδη αρκετές ερωτήσεις το ερώτημά μου είναι κάτι το οποίο με ρωτάνε συνεχώς στην εκλογική μου περιφέρεια. Εάν έχουμε φτάσει στον πάτο σε όλα τα κράτη-μέλη ή εάν πρέπει να περιμένουμε και χειρότερες ειδήσει. Δεδομένων των συζητήσεων που έχετε κάνει και του ρόλου σας στην Προεδρία, μπορείτε να με διαβεβαιώσετε πως από εδώ και πέρα τα πράγματα θα πάνε καλύτερα αντί για χειρότερα. Ευχαριστώ. Όπως είπα, πρώτη φορά σήμερα προείδρευσα. Τώρα αν αυτό με κάνει ειδικό για να μιλήσω για κάτι τέτοιο δεν το ξέρω, θα προσπαθήσω εν πάση Η διεθνής ε, κρίση υπάρχει εδώ και καιρό, μπορούμε να τρέξουμε στο 2008 με την γνωστή χρεοκοπία της ε, Lehman Brothers. Έχουμε δει πολλές χρεοκοπίες έκτοτε στο χρηματοπιστωτικό, στον τραπεζικό τομέα. Κανείς δεν μπορεί να αρνηθεί πως ε, έχουν γίνει πολλές προσπάθειες στην Ευρώπη και στο εξωτερικό και εκτός Ευρώπης για να διορθωθούν τα πράγματα. Οι συνεδριάσεις των G20, των G7, όλοι προσπαθούν να δουν την κατάσταση αυτή που προέκυψε από κάποιες αδυναμίες οι οποίες είναι εγγενείς στο σύστημα της ελεύθερης αγοράς και θεωρώ πως έχει γίνει πολλή δουλειά προς αυτή την κατεύθυνση. Θα ήθελα, ε, θεωρώ πως ε, έχουμε ήδη ξεκινήσει μια πορεία ε, προς το μέλλον. Πέρα από όλα τα υπόλοιπα δε, στην Ευρώπη είχαμε και την κρίση του ευρώ, οπότε τα πράγματα ήταν χειρότερα γιατί είχαμε ένα διπλό πρόβλημα. Τώρα, έχοντας όμως δει το τι συνέβη τους τελευταίους έξι μήνες, τις αποφάσεις οι οποίες ελήφθησαν, ακόμα και αν δούμε την απόφαση που ελήφθη πριν από δέκα μέρες από τους ε, αρχηγούς ε, κρατών, θεωρώ πως ε, έχουμε αντιμετωπίσει τα θεμελιώδη ζητήματα και αντιμετωπίζονται και αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Είμαι βέβαιος από αυτά που ξέρω από τις πληροφορίες που έχω στη διάθεσή μου πως τα πράγματα βελτιώνονται ε, ή τουλάχιστον είναι υπό έλεγχο. Και άρα μπορώ να πω πως είναι υπό έλεγχο. Πολλές συζητήσεις γίνονται για το πώς θα βελτιωθεί η κατάσταση. Η πρόεδρος. Ε, με συγχωρείτε, δεν μπορεί κάποιο να στέκεται στη μέση τη αίθουσα και να μην βλέπουν οι βουλευτέ που έκαναν την ερώτηση. Σα σας παρακαλώ, δεν είναι πράγματα αυτά. Έμα, αν στεκόταν μπροστά σου, είμαι σίγουρο, ε, Βέρνερ, όταν έκανε εσύ την ερώτηση, ότι δεν θα σου άρεσε. Ε, ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Μετά, μετά θα πάρετε το λόγο. Ο κύριο Σαρλή. Ε, είμαι αισιόδοξο. Θεωρώ πως ε, οδεύουμε προς μια έξοδο από την κρίση, από την κρίση του ευρώ, από την οικονομική κρίση. Υπομονή, θα βγούμε. Λυπούμε που σα διέκοψα, αλλά συνέβη και το πρωί. Μπενόβ να βοηθεί, μιλούσαν στους βουλευτές και μπλόκαραν τη θέα σε ευρωβουλευτές που κάθονταν πιο πίσω. Παρακαλώ λίγο μεγαλύτερη πειθαρχία. Τώρα θα ομαδοποιήσουμε τις ερωτήσεις, γιατί μας έχουν απομείνει μόνο 20, 25 λεπτά γιατί μέχρι τις 6.30 έχουμε την αίθουσα και τη διερμηνία. Ο Ζαν Πολ, ένα διαδικαστικό. Μέχρι τι ώρα κανονικά προβλέπεται η συνεδρίαση. Γιατί τροποποιήθηκε το αρχικό χρονοδιάγραμμα. Είχαμε πει αρχικά μία ώρα για την ε, συζήτηση. Αρχικά είχε προβλεφθεί για τρεις με τέσσερις. Αλλάξαμε βέβαια το πρόγραμμά μας για να έρθουμε αργότερα, αλλά νομίζω ότι η αυρότητα επιτάσσει μία ώρα διάρκεια. Ναι, αλλά μπορούμε να συνεχίσουμε μέχρι τις 6.30. Έχουμε την αίθουσα και τη διερμηνία μέχρι τις 6.30. Και ήταν και αρκετά μακροσκελής η ερωτήσεις. Ε, την ώρα την έχουμε ήδη ξεπεράσει, την αρχικά προβλεπόμενη. Ο κύριο Υπουργό όμω είπε ότι μπορεί να παραμείνει λίγο ακόμη, οπότε θα συνεχίσουμε μέχρι τις 6.30 αν δεν έχετε αντίρρηση και οι υπόλοιποι. Αλλά θα ομαδοποιήσω τώρα τις ερωτήσεις για να επιταχύνουμε κάπως τη συζήτηση. Αντολίν, Πρεζέντο, Ζάλμπα και Κάρας με τη σειρά που σας ανέφερα. Α, και ο Βέρνερ. Μετά. Όχι τώρα, Βέρνερ. Είσαι ο τρίτος. Ή μάλλον Άντολιν Παύλο και τρίτος ο Βέρνερ. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εκπρόσωπο της Κυπριακής Προεδρίας για την παρουσία του και την παρουσίαση των συστάσεων που μας έκανε για αυτό το εξάμεινο. Πιστεύω ότι το εξάμεινο είναι πολύ κατάλληλος μηχανισμός για την εμβάθυνση του οικονομικού συντονισμού στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εγώ θα αναφερθώ σε δύο συγκεκριμένα θέματα. Μία από τις χώρες που έλαβε τις περισσότερες συστάσεις, οκτώ τον αριθμό, ήταν η Ισπανία. Καμία άλλη χώρα δεν έχει λάβει τόσε συστάσει όσο η Ισπανία, από ό,τι ξέρω. Και δεύτερη ερώτηση για την Ευρωζώνη. Σε ό,τι αφορά την Ισπανία, θα μπορούσατε να μου επιβεβαιώσετε ότι όντως ε, έχουν γίνει δεκτές οι αλλαγές. Γιατί εγώ διαπίστωσα τρεις αλλαγές σε τρεις συστάσεις. Και κατά τη γνώμη μου είναι σωστές και οι τρεις αλλαγές, θετικές. Η μία, η πρώτη αλλαγή, αφορά την αύξηση της ε, ενημέρωσης και της ποιότητας των ε, δαπανών των διοικήσεων. Λογικό. Το δεύτερο είναι οι συντάξει, να προσαρμοστεί η ηλικία συνταξιοδότηση με το προσδόκιμο. Νομίζω ότι είναι καλύτερη η σύσταση αυτή αυτή που είχε προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και η τρίτη αλλαγή, ε, απασχολησιμότητα του ευάλωτου πληθυσμού και των ε, οικογενειών με χαμηλά εισοδήματα. Ωραία αυτά. Επίσης παραχωρήθηκε ένα χρόνος ακόμη για την Ισπανία για να κάνει την προσαρμογή. Νομίζω ότι είναι λογική αυτή η παράταση. Και επίση η φορολογική εξυγίανση θα πρέπει να γίνει με ευφύ τρόπο. Βέβαια, πριν από τρει μήνες όταν υπευλήθησαν οι προπολογισμοί από την Ισπανική κυβέρνηση, προπολογισμοί που αναφερόταν σε έλλειμμα 5,8% και τελικά το Συμβούλιο είπε ότι θα πρέπει να είναι γύρω στο 5,3%. Τώρα δέχτηκε το 6,3%. Αυτή είναι η επίκρισή μου. Με παρόμοιες πληροφορίες με αυτές που έχουμε τώρα. Ίσως αυτό θα πρέπει να το θέσουμε στα αρνητικά του Συμβουλίου, στα μείον, γιατί σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα το Συμβούλιο άλλαξε την προσέγγιση του και το κριτήριο. Ήδη από, από την αρχή θα μπορούσε να έχει υιοθετήσει το πιο ελαστικό και το πιο λογικό κριτήριο. Η δεύτερη ερώτηση αφορά την ειδική προθεσμία για ένα πολιετές ε, ε, πρόγραμμα για δύο χρόνια. Είπαμε τέλη Ιουλίου. Και ε, προβλέφθηκε η περίοδος ελέγχου για τρεις μήνες. Θα ήθελα να πω ότι είμαι υπέρ και των συστάσεων για την Ευρωζώνη αλλά και εκεί υπάρχει μια παράληψη. Κρίμα να μην υπάρχουν προθεσμίες στις συστάσεις για την Ευρωζώνη, γιατί όταν μπαίνουν προθεσμίες για τις χώρες στις συστάσεις, καλό θα είναι να μπαίνουν προθεσμίες και στις συστάσεις για την Ευρωζώνη. Άλλωστε και στη Συμφωνία του Συμβουλίου έχουμε κάποιες ημερομηνίες αναφοράς. Καλό θα ήταν και προθεσμίες να είχε περιλάβει το Συμβούλιο στις συστάσεις του φεύγουν στο μεταξύ κάποιοι που θέλουν να υποβάλουν ερωτήσει εξαιτία του αργού ρυθμού. Ο Παύλο έφυγε στο μεταξύ η Άστριτ και η Άννη και μετά θα ακούσουμε τι απαντήσει από τον Υπουργό. Ο Παύλο. Ευχαριστώ Σάρον. Αγαπητέ κύριε Υπουργέ, θα θέλαμε και εμεί να σα ευχαριστήσουμε για την παρουσία σα εδώ και να αναφερθώ σε ένα πολύ συγκεκριμένο θέμα, την Τραπεζική Ένωση. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ήταν ανέκαθεν υπέρμαχο αυτού του θέματος και χαιρόμαστε που και το Συμβούλιο η τελευταία μάλιστα διάσκεψη κορυφή τη προηγούμενη ε, Πέμπτης ε, έφτασε, κατέληξε σε συμφωνία για το θέμα αυτό. Επιτέλους ε, ανακάλυψαν τα πλεονεκτήματα αυτή της πρόταση τη Τραπεζική Ένωσης. Το Συμβούλιο έδωσε ξεκάθαρη εντολή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να καταρτήσει πρόταση για το θέμα αυτό με συγκεκριμένη προθεσμία. Κάποια μέλη όμω του Συμβουλίου μίλησαν για εύλογε προθεσμίες ε, σε ό,τι αφορά την εφαρμογή. Άλλα μέλη του Συμβουλίου όμως ε, είπαν ότι μπορούν να καθυστερήσουν και χρόνια ολόκληρα μέχρι να φτάσουμε στη υλοποίηση αυτής της Τραπεζικής Ένωσης. Εσείς ε, ως Προεδρεύον του ΕΚΟΦΗΝ, τι γνώμη έχετε. Πιστεύετε ε, ότι θα επικρατήσουν οι πιο αισιόδοξε ή οι πιο απεσιόδοξε προτάσει ό,τι αφορά την ε, προθεσμία για την εφαρμογή τη Τραπεζική Ένωση. Ευχαριστώ, Σάρων. Κύριε Υπουργέ, κύριε Σάλη, δεν σκοπεύω να σας φέρω σε δύσκολη θέση και να κάνω ερώτηση για την Ελλάδα. Η σύσταση για την Ελλάδα είναι σύντομη. Λέει απλά εφαρμογή του προγράμματος. Και όπως ξέρετε αυτό ακριβώς σκοπεύει να κάνει η νέα κυβέρνηση και ο νέος υπουργό Οικονομικών. Θέλω μόνο να επισημάνω πως είναι αντιπαραγωγικό να θεωρείται η χώρα, οποιαδήποτε χώρα, ε, υπεύθυνη για όλα τα κακά του κόσμου ή ως ένας δαίμονας ε, εντός της Ευρωζώνης και του δουλεχθέντος θέλω να επανέλθω στα σχόλια της συναδέλφου μου, της, συναδέλφου Ελίζας για, τις, ε, για τη χώρα της και στις δικές παρατηρήσεις για την Κύπρο. Να ένα θέμα είναι το ζήτημα της αλληλεξάρτησης. Ε, δεν ε, υπάρχει καμία αμφιβολία πως το κούρεμα παραδείγματος χάρη των ελληνικών ομολόγων και η έκθεση των κυπριακών τραπεζών στην Ελλάδα είχε τεράστιο κόστος, αλλά υπήρχαν και προβλήματα δημοσιονομικά, αλλά η αλληλεξάρτηση είναι ε, ένα θέμα και η συνταγή και το αν αυτή είναι σωστή είναι κάτι άλλο. Και θα ήθελα να σας ε, ρωτήσω λαμβάνοντας υπόψη ε, τις προτάσεις που έγιναν από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την Επιτροπή μας, η Ελίζα ανέφερε τις εξοδηγίες. Εγώ αναφέρομαι στο λεγόμενο πακέτο των δύο οδηγιών, τους νέους ε, τους νέους κανονισμούς για ενισχυμένη επιτήρηση Ε, πως οι χώρες οι οποίες ε, λοιπόν είναι υπό το καθεστώς αυτό του προγράμματος ε, προσαρμογής πρέπει να μπορέσουν να επιδείξουν μια κάποια ευελιξία δηλαδή να ληφθεί υπόψη, να ληφθούν υπόψη τυχόν αποκλήσεις από τους στόχους, μακροοικονομικές ανισορροπίες ή αποκλήσεις ε, που είναι οφείλονται σε λόγους πέρα από τη θέληση και την ε, δυνατότητα των κρατών μελών ή μεγαλύτερη ευελιξία για να είναι πιο αποτελεσματικά. Αυτή ήταν η πρόταση του Κοινοβουλίου. Θα ήθελα να σας ρωτήσω εάν ε, υποστηρίζετε μια τέτοια προσέγγιση. Ευχαριστώ. Υπάρχει ο τριμερής διάλογος, λέει η Πρόεδρος, για αυτό το θέμα αύριο και ο Ανδρέας επίσης θα διαπραγματευτεί εκπροσωπώντα την Προεδρία. Αλλά δεν νομίζω πως εδώ είναι η κατάλληλη στιγμή για αυτό το διάλογο. Μπορείτε λοιπόν να αποκαλύψετε και να παραχωρήσετε στο Κοινοβούλιο ό,τι θέλετε τώρα. Regarding the first question, which, um... Για το πρώτο ε, ερώτημα για την Ισπανία και τις οχτώ συστάσεις που έγιναν ειδικά προς την Ισπανία. Νομίζω πως οι συστάσεις ήταν πραγματικά πολύ κέρυες και ο Υπουργό Οικονομικών Λουίς σήμερα ενημέρωσε το ΕΚΟΦΗΝ και χθε το βράδυ το Eurogroup για την ε, αποδοχή των συστάσεων ως ε, απαραίτητη προϋπόψη, αλλά όχι ακριβώς με τη μορφή που έχουν, ακριβώς γιατί αυτές οι συστάσεις ε, απαντήθηκαν. Για τον λόγο αυτό η Ισπανία όχι μόνο έλαβε την βοήθεια που ήθελε για ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών της, αλλά και μια παράταση για ένα έτος για την εφαρμογή της μείωσης του ελλείμματος του προπολογισμού από το 6,3 ή πόσο είναι τέλος πάντων στο, στο 2% μέχρι το 2014 αυτό. Οπότε ε, τέλος δεν μπορώ να πω σε λεπτομέρειες αλλά η συνολική αυτή προσέγγιση των συστάσεων είχε κάποια ουσία ε, δηλαδή υπήρχε κάποια ουσία και απαντώντα σε αυτό το Eurogroup και το ECOFIN σήμερα ε, ενέκρινε όλα τα αιτήματα ε, βοήθειας της Ισπανίας. Οπότε βλέπετε πως η Ευρώπη είναι, είναι στο πλευρό της, υπάρχουν τα μέσα, υπάρχουν τα κονδύλια για να βοηθήσουμε να τα Είναι λοιπόν μια αμφίδρομη διαδικασία, γι' αυτό αναφέρθηκα και στην Ελλάδα υπό την εντύπωση η Ελλάδα έχει πρόβλημα, το ξέρουμε όλοι, αλλά αναφέρθηκα στην έννοια της αλληλεγγύης. Πρέπει να επιδείξουμε αλληλεγγύη προς την Ελλάδα. Ταυτόχρονα όμως, όπως είπα, πρέπει να αναγνωριστούν και οι υποχρεώσεις. Και μάλιστα, μιλώντας σήμερα στον νέο Υπουργό Οικονομικών της Ελλάδας, τον κύριο Στρονάρα, και ο ίδιος είπε χθε το βράδυ στο Eurogroup επιβεβαίωσε πως η Ελλάδα θα εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της. Ε, ήταν απόλυτος αυτό. Και είναι πάρα πολύ θετικό αυτό και είναι ένα μήνυμα ακριβώς πως αυτά πάνε μαζί. Υποχρεώσει και αλληλεγγύη. Όσον αφορά την Τραπεζική Ένωση, θεωρώ πως αυτό είναι ένα νέο θέμα που προέκυψε τώρα τελευταία, πρέπει να γίνει πολύ δουλειά ακόμα προς αυτή την κατεύθυνση, είναι μία από τις προτεραιότητες του ΕΚΟΦΗΝ και θα το εξάσουμε και θεωρώ πως πάρα πολύ σύντομα θα έχουμε μία πρόταση από την Κομισιόν. Αλλά μιλώντας ναι, για κάτι στο οποίο αναφέρθηκα πριν για την ενιαία εποπτική αρχή που είναι ένα συστατικό μέρος μιας ε, τραπεζικής ένωσης, ένα προαπαιτούμενο, ε, είναι ένα κομμάτι το οποίο όταν θα το έχουμε θα δούμε αυτό το οποίο ε, προανέφερα πριν, πως θα βλέπουμε πλέον μία διέξοδο, θα επανέρχεται η εμπιστοσύνη, οι χρηματαγορές θα βασίζονται σε δεδομένα και το τραπεζικό σύστημα που είναι τόσο σημαντικό βεβαίως, ε, για να μπορέσουμε να στηρίξουμε την οικονομία, αλλά και όσον αφορά και το δημόσιο χρέος, ε, πράγματα τα οποία είναι αλληλένδετα. Did Μήπως θα θέλετε να μας πείτε ότι μας δίνετε ό,τι διεκδικούσαμε για το διπλό πακέτο. Δεν ξέρω αν θέλετε να προσθέσετε κάτι και για το πακέτο των δύο οδηγιών, το δίπτυχο. Ας μην προδικάζουμε την αυριανή πολύ ενδιαφέρουσα από ό,τι φαντάζομαι συζήτηση. Αυτά τα θέματα θα συζητηθούν αύριο. Ε, δεν μα ευνηδιάζετε, δεν μα εκπλήσετε. Ελπίζω ότι θα σημειωθεί πάντω πρόοδο αύριο. Ευχαριστώ πολύ και ζητώ συγγνώμη σε όσου δεν πρόλαβα να θέσουν ερωτήσει και χρειάστηκε να φύγουν. Αλλά φταίνουν οι συντονιστέ που έθεσαν πολύ μακροσκελείς ερωτήσεις και δεν έμεινε χρόνος για τους υπόλοιπους. Πάντως σας ευχαριστούμε κύριε Υπουργέ που βρήκατε το χρόνο και ήρθατε, γιατί ξέρουμε είναι δύσκολο να αφήνετε το κοφί στη μέση. Πάντως, σε περίπτωση που δεν το ξέρετε, η επόμενη μα συνεδρίαση θα γίνει στις 3 Σεπτεμβρίου, στις 3 ώρα το απόγευμα. Σας ευχαριστώ.